στην κυρία Σίπελ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, του κύριε Επίτροπε, Ρέντινγκ, κύριε συνάδελφοι. Ακριβώς αυτές τις ε, μέρες, τις εβδομάδες, τους μήνες είναι σημαντικό να τονίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι παραπάνω από μια αγορά. Είναι μια κοινότητα αξιών και αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται ακριβώς σε δύσκολους καιρούς όπου θα πρέπει να δεχτεί ισχυρή σε όλους τους τομείς της πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη βασίζονται στις κοινέ αρχές ελευθερίας, δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Και ένα αναπόσπαστο τμήμα της, του κράτους δικαίου σε σχέση με τις ε, σπιτικέ διαδικασίε είναι ε, ότι ο κατηγορούμενος θεωρείται καταρχήν αθώος. Μετά την οδηγία για την μετάφραση και διερμηνία, η νέα οδηγία για την ενημέρωση ε, στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών είναι ένα σημαντικό βήμα, ούτως ώστε όλοι οι κατηγορούμενοι να τη χάνουν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίκαιες δίκες. Κάτι τέτοιο αυξάνει την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών στο κράτος δικαίου και στην δικαιοσύνη και η αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων προωθείται επίσης. Ο, το μεμονό άτομο μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μόνο εάν τα γνωρίζει και για μια δίκαιη ε, δίκη είναι σημαντικό να γνωρίζει κανένα τα δικαιώματά του, να γνωρίζει τι του προστάτεται και αν καταπατούν τα δικαιώματα αυτά διακυβεύεται η δίκαιη ε, εξέλιξη της δίκης. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δικαιοσύνη συγκεντρώνονται στην καλύτερη συνεργασία. Η νέα διαδικασία όμως έχει σαν στόχο τους πολίτες και τα δικαιώματά τους προβλέπει οι αστυνομικές αρχές και οι δημόσιοι κατήγοροι και οι εισαγγελείς να ενημερώνουν τους ε, κατηγορούμενους με απλά λόγια για τα δικαιώματά τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει επίσης το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης και το δικαίωμα να δουν το δικαστή αμέσως μετά την σύλληψη. Ε, ε, το Κοινοβούλιο θέλει να διευρύνει τα δικαιώματα των κατηγορών, παραδείγματος χάρη ιατρική περίθαλψη, επαφή με τους ε, συγγενείς και το δικαίωμα άρνησης δήλωσης. Έξι λεπτά έχω πρόεδρε. Κανένας δεν ξέρει πόσο χρόνο παραμένει ένας κατηγορούμενος σε προδικαστική φυλάκιση και γι' αυτό είναι σωστό να γνωρίζει τα δικαιώματά του και να έχει και πρόσβαση σε ελαφρυντικά στοιχεία. Ο κατηγορούμενος δεν πρέπει να είναι αντικείμενο της διαδικασίας, θα πρέπει να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία αυτή. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν τώρα να υιοθετήσουν την οδηγία αυτή και να την εφαρμόσουν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές που πρόθεσαν την έκθεση αυτή με καλή συνεργασία. Είναι σημαντικό τώρα πια το Συμβούλιο και η Κομισιόν να προωθήσουν τα περαιτέρω μέτρα της οδηγίας αυτής να ολοκληρώσουν το γρηγορότερο δυνατόν ούτως ώστε να υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πρότιμα και δίκαιες δικαστικές διαδικασίες. Ευχαριστώ. Thank you very much. That was your minutes. Uh, Ευχαριστώ. Αυτά ήταν τα έξι λεπτά. Τέσσερα τώρα, δύο στο τέλος, όλα μαζί. Η κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά που έκανε και για τον αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής των ε, διαπραγματεύσεων. Αυτό επέτρεψε μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Θα ήθελα επίσης να επενέσω το ρόλο του κύριου Άλμπρεχτ που συνέταξε για την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων το κείμενο και για το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν και όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εν γέννη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι συμβάλλατε στο να διατηρηθεί το επίπεδο των φιλοδοξιών της Προτάσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίως κάτι που πιστεύω ότι είναι σημαντικότατο για τους πολίτες μας. Το τη χάρτα των δικαιωμάτων που έπρεπε να παραμείνει στο τελικό κείμενο κατάλογος δικαιωμάτων και τη στιγμή που αρχίζουν να ισχύουν αυτά τα δικαιώματα. Καλωσορίζω το γεγονός ότι και συμπροματικά δικαιώματα προστατεύθησαν στον κατάλογο των δικαιωμάτων, κυρίως το δικαίωμα να μένει κανείς σιωπηλός. Να σιωπά κανείς που δείχνει κανείς ότι είναι πολύ καλό ότι το Κοινοβούλιο έχει δυνατότητα συναποφάσεως, διότι το Κοινοβούλιο προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων. Το δικαίωμα πληροφόρησης και ενημέρωσης σε διάφορες ποινικέ ε, υποθέσεις είναι ένα τμήμα του δικού χάρτη για ε, τα διαδικαστικά δικαιώματα και η εφαρμογή αυτού του δικού χάρτη ε, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για μένα. Τώρα, το δικαίωμα πληροφόρησης και ο κατάλογος δικαιωμάτων είναι το δεύτερο μέτρο που υιοθετήθηκε το δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνίας ήδη έχει υιοθετηθεί. Άρα κάνουμε Σημειώνουμε πολύ γρήγορη πρόοδο και πιστεύω ότι αυτό είναι καλό για την Ευρώπη των πολιτών και για τα δικαιώματα των πολιτών. Σε κάποια κράτη-μέλη μου ετέθη το ερώτημα, βλέπετε, ή το κάνετε αυτό, με ρωτάνε. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι τα συνηθισμένα δικαιώματα που απολαμβάνει ο καθένας. Δυστυχώς, σε κάποια κράτη-μέλη κάποιος μπορεί να προσαχθεί σε δίκη και να μην ξέρει ότι έχει το δικαίωμα δικηγόρου ή διερμηνέα. Έχουμε ακούσει και περιπτώσεις όπου υπάρχουν άνθρωποι που δικάστηκαν και δεν γνώριζαν ή δεν κατάλαβαν ποια ήταν η κατηγορία εναντίον τους. Έτσι λοιπόν, χάρη στο μέτρο αυτό, οι κατηγορούμενοι θα έχουν ένα έγγραφο δικαιωμάτων σε μια γλώσσα κατανοητή σε αυτούς και θα είναι βέβαιο ότι θα έχουν επαρκή ενημέρωση για τις κατηγορίες που απαγγέλλονται εναντίον. Αυτό είναι σημαντικό στη σημερινή Ευρώπη όπου εκατομμύρια άνθρωποι ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης και μετακινούνται σε άλλα κράτη-μέλη για εργασία, για σπουδές ή και για την ε, συνταξιοδότησή τους. Είναι σημαντικό εάν βρεθούν ε, λεγμένοι σε κάποια ποινική διαδικασία να προστατεύονται τα, δικαιώματά τους και το Κοινοβούλιο έχει βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση επιπλέον. Το μέτρο αυτό θα ε, παίξει σημαντικό ρόλο στην ε, προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών, που και αυτό είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της δικατικής συνεργασίας ε, γιατί χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Αυτά είναι λοιπόν τα μέσα της ε, αμοιβαίας αναγνώρισης που δημιουργούμε για τους Ευρωπαίους πολίτες και ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου που το καθιστούν δυνατό. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Τώρα έχει το λόγο εξ της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για 1,5 λεπτό ο συνάδελφος κύριος Άλμπρεχτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, εισηγητής της Νομικής Επιτροπής θα ήθελα ε, καταρχήν να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου εμείς ως Νομική Επιτροπή είχαμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε με τις δικές μας προτάσεις ε, στη διαδικασία. Και τα συγχαρητήριά μου απευθύνονται επίσης και στην επίτροπο που θέτει ένα νέο λίθο στο οικοδόμα για τη δημιουργία κοινών ε, προδιαγραφών. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτών των κοινών προδιαγραφών. Και είναι σημαντικό και για τους πολίτες, γιατί μόνο ενήμεροι πολίτες που γνωρίζουν τα δικαιώματά τους μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των δικαιωμάτων και γι' αυτό αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία θα μπορούμε να ξεπίσουμε μελλοντικά ως Ευρωπαίοι πολίτες. Έχω το βλέμμα μου λοιπόν στραμμένο προς το μέλλον και ελπίζω ότι σύντομα θα γίνουν και τα περαιτέρω βήματα που αφορούν την ε, δυνατότητα προσφυγής ε, σε δικηγόρο, όπου εγώ ως κοιόδης συγητής στην Επιτροπή Ιστορικών Υποθέσεων πρόκειται να παρακολουθήσω αυτή τη διαδικασία, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να καλέσω και τις χώρες μέλη εδώ να ξεπεράσουν τις αντιστάσεις απέναντι σε επιμέρους διατάξεις και να κινηθούν προς την κοινή οδό για τη δημιουργία αυτών των κοινών ε, προϋποθέσεων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Άλμπρεχτ και τώρα θα περάσουμε στον κύριο των ομιλητών που παρεμβαίνουν εξ ονόματος των διαφόρων κοινοβουλευτικών ομάδων. Καταρχήν για δυόμιση λεπτά εξ ονόματος του ΕΛΚ η συνάδελφος κυρία Ελένα Αντωνέσκου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία για τους κατηγορούμενους είναι πραγματικά εκ των ουκάνευ. Το να, το να έχουν ε, οι άνθρωποι αυτοί πληροφορίες είναι προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανεξάρτητα από την κατηγορία που τον βαρύνει και ανεξάρτητα από τα ε, επιβαρυντικά στοιχεία τα οποία ε, υπάρχουν εναντίον του, έχει κάθε δικαίωμα να δεχτεί αυτήν την πληροφορία. Αυτή τη στιγμή διαφέρουν οι διαδικασίες από χώρα σε χώρα ε, και επομένως ε, ε, δεν υπάρχει μία ισοδίκαιη αντιμετώπιση. Επίσης πολύ συχνά ε, είτε δεν είναι δίκαιες οι δίκες, είτε δεν ε, προχωρούν τελικά οι διαδικασίες ε, ή αργούν υπερβολικά. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει της, σύμβαση, της συνθήκης, της σύμβασης συγγνώμη, για τις θεμελιώδες ελευθερίες δεν ε, αποτελεί ικανοποιητικό βαθμό προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, χρειάζεται ε, κοινοτική δράση. Τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς διευκόλυνση της δικαϊκής συνεργασίας βασίζονται στην αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης των αποφάσεων και στην αυτόματη αναγνώριση σημαντικών κανόνων. Πράγμα απολύτως θεμελιώδες για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και μεταξύ των δικαστών. Ε, όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει τελικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε επομένως καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές ε, για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν, καθώς επίσης ε, να ευχαριστήσω και την Επίτροπο, η οποία έχει στρατευτεί έτσι ώστε να επιτύχει αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντωνέσκου. Τώρα Παρακαλώ, κυρία Αντωνέσκου. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Και πάλι θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι συνάδελφοι διερμηνείς ε, μου είπαν ότι μιλάτε με μεγάλη ταχύτητα. Ε, θα ήθελα να σας επισημάνω και πάλι ότι υπάρχει μία ένδειξη στις οθόνες σας που δείχνει την υπερβολική ταχύτητα. Όταν δείτε αυτή την ένδειξη, παρακαλώ να επιβραδύνετε το ρυθμό ομιλία σας για να μπορείτε να μεταφραστείτε σε όλες τις γλώσσες. Ε, κυρίως όταν διαβάζετε ένα κείμενο θα πρέπει πραγματικά να μετράσετε το ρυθμό ομιλία σας. Όταν δείτε αυτή την ένδειξη, όταν ανάβει η ένδειξη στην οθόνη σας, ε, παρακαλώ να καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει διερμηνία λόγω της υπερβολικής ταχύτητας. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντωνέσκο για την κατανόησή σας. Και τώρα εκ μέρους των συναδέλφων σοσιαλιστών έχει το λόγο για 1,5 λεπτό η κυρία Μόνικα Πλασίκοβα Μπένοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Και κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο χάρτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει ότι ένα βασικό δικαίωμα του κατηγορουμένου είναι το δικαίωμα επαφής με το δικηγόρο, διερμηνίας, μετάφρασης, ενημέρωσης και της ε, ενημέρωσης για την διαδικασία. Η πρόταση αυτή επικεντρώνεται στη βελτίωση των δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων και κυρίως στην ενημέρωσή τους. Καλύπτει επίσης περιπτώσεις, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος συλλαμβάνεται επί τη βάση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αυτά είναι ελάχιστα πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα πρέπει να διευκολύνουν την εφαρμογή της αμοιβαία συνεργασίας και δικαστηρίων και κρατών μελών. Συμφωνώ με τη θέση της Νομικής Επιτροπής, η οποία ε, αναφέρει ότι στο σχέδιο που ε, προωθούμε η προσέγγιση είναι κατακαιρματισμένη. Εδώ έχουμε ένα δεύτερο μέτρο που και ως εκ τούτου η πρόταση της Επιτροπής αποκλεί εν μέρη κάποια δικαιώματα και έχει μόνο το μισό ε, ε, σύμφωνο των δικαιωμάτων. Δηλαδή έχει το δικαίωμα του δικηγόρου και το, ε, αναφέρονται τα δικαιώματα αυτών που είναι βάλωτα άτομα. Θα πρέπει να τροποποιηθούν και με τα επιπλέον δικαιώματα κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μόνικα. Τώρα έχει εκ μέρου των φιλελευθέρων για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Σάρα ε, Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που μας οδήγησε σε επιτυχημένο συμπέρασμα. Πάντοτε είναι ευπρόσδεκτη η ε, υποστήριξη της Αντιπροέδρου κυρίας Ρέντινγκ Οπωσδήποτε κάποιος ο οποίος ε, υφίσταται ανάκριση ε, βρίσκεται σε ευάλωτη θέση. Η ποιότητα των πληροφοριών που, προσφέρεται συνήθως δεν είναι καλή. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από το γεγονός ότι κάποιος είναι ξένος ή δεν μιλάει τη γλώσσα. Υπάρχει διάκραση γιατί πρέπει κανείς ε, ας πούμε για να του δοθεί δικαίωμα αναστολής να κάνει τις απαραίτητες νομικές κινήσεις και να γνωρίζει τα δικαιώματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει λοιπόν οι πληροφορίε αυτέ να παρέχονται το ταχύτερο δυνατόν, μόλι ενημερώνεται κάποιο για το καθεστώ του υπόπτου. Δεν θα πρέπει κανεί να αφήνεται να ψήνεται σε ένα κελί τη αστυνομία, αστυνομικού τμήματο, χωρί να μπορεί να έχει βοήθεια από δικηγόρο. Επίση, ο δικηγόρος και ο κατηγορούμενος πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο από, την, ε, από τις διοκτικές αρχές. Όπως και η κυρία Ρέντινγκ συμφωνώ ότι το δικαίωμα του να παραμείνει κανείς σιωπηλός είναι ένα θετικό δικαίωμα. Όπως επίσης υπάρχει και το δικαίωμα στην διερμηνή και τη μετάφραση. Ελπίζω ότι θα λάβουμε μέρος και το τρίτο μέτρο στην πρόσβαση στι νομικές συμβουλές. Και έχουμε καλό ιστορικό και η χώρα μου πρέπει να εμπλακεί απόλυτα. Βεβαίω, έχουμε ε, καθυστερήσει πολύ στην ε, ενίσχυση ε, των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων σε σχέση με την ενίσχυση των δικαιωμάτων της δίωξης. Έτσι λοιπόν θα πρέπει οι καταστάσεις που έχουμε γνωρίσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης να περάσουν στο παρελθόν Τώρα εξ ονόματος των Ευρωπαίων Μεταρρυθμιστών για ένα λεπτό έχει το λόγο ο συνάδελφος κύριος Βολτσεχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφερόμαστε εδώ σε μια οδηγία η οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμη η οποία επίσης καταδεικνύει ότι χρειάζεται διαφάνεια στη διαδικασία ε, όσον αφορά το δικαίωμα υπεράσπισης. Το δε δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μονάχα εάν ο κατηγορούμενος έχει όλα τα στοιχεία, τα αποδεικτικά, τα τεκμήρια, τα οποία ε, έχουν ιδιοκτικές αρχές και βάσει των οποίων ε, τον κατηγορούν. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό μέχρι τώρα δεν γίνεται. Η δυσκολία δε γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν κάποιος βρίσκεται σε ξένη χώρα της οποίας τη γλώσσα δεν μιλάει αυτές τις περιπτώσεις ε, θα πρέπει να στραφούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Δέχομαι όλες τις προτάσεις της οδηγίας, αλλά έχω κάποιες αμφιβολίες όσον αφορά την υλοποίηση. Ε, δεν ξέρω εάν θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις, ε, γιατί τα ζητήματα δικαιοσύνης είναι περίπλοκα. Αναρωτιόμαστε εάν η οδηγία αυτή θα μπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα ε, ε, όπου και οι προσφυγές να είναι δυνατές. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Εξ ονόματος της Ευρώπης Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, ο συνάδελφος Τζέραρ Μπάρτον ένα λεπτό. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνεται το δικαίωμα ε, ενημέρωσης του συλληφθέντος. Ε, και ε, στην περίπτωση γραπτής διαδικασίας ε, θα μιλάμε για μια σύντομη επιστολή. Αλλά βεβαίως εάν δεν υπάρχει σωστή συμπλήρωση της φόρμας, του, του αιτήματο, ε, τότε το δικαστήριο σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν θα έχει ε, μεγάλες επιλογές. Το σημαντικό είναι όλες αυτές οι διαδικασίες να κινηθούν όχι από τη στιγμή που θα υπάρξει καταδίκη, αλλά στη διάρκεια της προδικαστικής διαδικασίας. Στην περίπτωση της δική μου εκλογικής περιφέρειας έχω πολλέ περιπτώσει τις οποίες μπορώ να σας ε, υποβάλλω ε, και κατά την, ε, και σε αυτές τις περιπτώσεις όλες δεν έχει υπάρξει σωστή ενημέρωση με αποτέλεσμα ο δικαστής να μην έχει άλλη λύση παρά την καταδίκη του ατόμου. Πρόεδρος, εξο... Εξαντλήσαμε το κατάλογο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Τώρα θα μιλήσουν οι αγορητές που παίρνουν το λόγο ατομικά. Για ε, πρώτος ο κύριος Μπαλτασέρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Παρότι ε, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν ε, να αντιμετωπίζουν ισοδίκαια τις, δικαστικέ τα... δικαστικές διαδικασίες των ατόμων, γνωρίζομαι ότι οι ποινικέ διαδικασίες ποικίλουν ε, έντονα. Ε, σε μερικές περιπτώσεις μονάχα προφορικά ενημερώνονται περί των διαδικαστικών ε, οι κατηγορούμενοι. Άλλοι, ε, οι άλλες χώρες δίνουν γραπτές περίπλοκες τεχνικές πληροφορίες μονάχα γραπτά ε, και μετά από αίτημα ε, των ε, ενδιαφερομένων. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κάθε χρόνο έχουμε 8 εκατομμύρια περιπτώσεων θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Επομένως, συμμερίζομαι πλήρως το πνεύμα αυτής της οδηγίας. Κυρίως δε στο σημείο που αναφέρει ότι θα πρέπει να δίδονται στον κρατούμενο πριν από την αρχή της δομικής διαδικασίας ε, όλες οι πληροφορίες ε, σχετικά ε, με το υλικό της δικογραφίας, την ενημέρωση του δικηγόρου, ενημέρωση σχετικά με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας γενικότερα. Επίσης θα πρέπει να έχει πλήρη δικαίωμα ενημέρωση όσον αφορά ε, όλα τα στοιχεία τα οποία θεωρούνται επιβαρυντικά θα πρέπει να έχει δυνατότητα μετάφρασης ερμηνείας έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός περί τίνος πρόκειται και να οργανώσει μαζί με τον ε, δικηγόρο του την καλύτερη δυνατή ε, υποστηρικτική γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον και του συσκιώδεις που έχουν συνεργαστεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια καλή η, ε, ε, διαδικασία. Αγαπητέ συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος, και ο τόνος της φωνής σας και ο, ε, ο ρυθμός σας είναι το όνειρο του κάθε διερμηνέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, νομίζω, ελπίζω δηλαδή ότι όλοι θα μιλάνε με αυτόν τον τρόπο. Έχει το λόγο για 1,5 λεπτό η συνάδελφος κυρία Μπλίνκεβιτσιουτέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση. Πραγματικά μιλάμε για ένα σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση του να εξασφαλιστούν κοινά ελάχιστα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα στην ενημέρωση κατά την ποινική διαδικασία. Δεν αρκεί να γνωρίζει κανείς τα δικαιώματά του. Σημαντικό είναι να γίνονται σεβαστά και να ασκούνται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί αν όχι μπορούν να τεθούν σε κίνδυνο οι ποινικέ διαδικασίες και να οδηγήσουν σε κακοδικία. ω εκ τούτου τα μέτρα αυτά επιδιώκουν την επίτευξη, την διεξαγωγή μιας δίκαιας δίκης και στη χώρα προέλευση αλλά και σε οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαίωμα ε, για ε, προσφυγή σε δικηγόρο ή σε διερμηνία και μετάφραση για να εξασφαλιστεί η δίκαιη δίκη και το δικαίωμα υπεράσπισης στα κράτη-μέλη πρέπει οι υποπτοί και οι κατηγορούμενοι να, έχουν τη δυνατότητα ε, πρόσβασης πρόσβαση ε, πληροφοριών για τα αίτια της... Ε, των κατηγοριών. Δεν θα πρέπει οι πληροφορίες να περιορίζονται στο δικαίωμα της νομικής βοήθειας και συμβουλής αλλά τη δυνατότητα να έχει κανείς επαφή με τα μέλη της οικογένειάς του, συγγενείς, τους ή τις προξενικές αρχές έχει το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Άξελ Φως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε Ρέντινγκ. Καταρχήν θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το αποτέλεσμα της εργασίας της Μπίργκετ Ζίπελ ε, και ε, με βρίσκει απολύτως ε, σύμφωνο με την ε, πρόταση να διατυπωθούν ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την ενημέρωση των κρατουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ευθύ εξ εξαρχή θεώρησα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και θα ήθελα σε εκ τούτου να ευχαριστήσω ιδιαίτερος την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ και να τη συγχαρώ. Ε, ιδιαίτερο σημαντικό στα πλαίσια της διαδικασίας ήταν ε, για μένα τα δικαιώματα του υπόπτου, ιδιαίτερα το δικαίωμα της σιωπής να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις όπως ε, συμβαίνει σε ορισμένες ε, χώρες μέλη. Αυτό σήμερα εξασφαλίζεται και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό και ε, στην ε, συζήτηση για την έκθεση αυτή έγινε προφανές ότι σε πολλές χώρες μέλη δεν υπάρχει νομική δέσμευση να ενημερώνεται ο κρατούμενος για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν μόνο σε 10 χώρες ε, μέλη πρέπει να ενημερώνεται εγγράφος ο κατηγορούμενος για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν και ε, μόνο σε τρεις χώρες, ε, και σε τρεις χώρες δεν υπάρχει καθόλου δυνατότητα πρόσβασης στη δικογραφία. Αν δούμε τι γίνεται στη Γαλλία όσον αφορά τη λεγόμενη garde à vue, εδώ διαπιστώνουμε ότι κατά την πρώτη φάση της κράτησης δεν υπάρχει δυνατότητα ε, αρρωγής από δικηγόρο. Έτσι διαπιστώνουμε την ανάγκη να υπάρξει μια εξομοίωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συν το χρόνο, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και σε άλλα συστήματα δικαιοσύνης, ούτως ώστε να υπάρξει μια βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης χωρίς να έχουμε πετύχει ένα επαρκές επίπεδο δεν είναι δυνατόν να λάβουμε μέτρα όπως για παράδειγμα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη και να το προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι με την έκθεση αυτή κάνουμε ένα ε, βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φως. Τώρα έχει το λόγο για 1,5 λεπτό η κυρία Κάρμεν Ρομέρο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πρωτίστως να αναγνωρίσω την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ και στην Επιτροπή την προσπάθεια που κατέβαλε ώστε αυτή η δέσμη των δικονομικών εγγυήσεων να γίνει πιο ευέλικτη και να προχωρήσει. Ε, και δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί ε, ο δικός χάρτης. Ε, πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό ιδιαίτερα σημαντική αυτή η πρόταση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πίρκετ Τσίπελ για την προσπάθεια που έκανε για να θεσπίσει αυτή την πρόταση οδηγίε ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι ουσιαστικά όσον αφορά τον κατηγορούμενο για την, ε, με τι κατηγορίες βαρύνεται για παράδειγμα και επίσης το δικαίωμα της σιωπής καθώς και το δικαίωμα να αγνωρίζει τα αδικήματα για τα οποία κρατείται. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω περισσότερο σε αυτή την παρέμβαση είναι η συζήτηση που έγινε σε σχέση με το δικαίωμα της, στη μετάφραση και τη διερμηνία καθώς και το δικαίωμα της νομικής αρρωγής για έναν κατηγορούμενο. Πότε θα πρέπει να γίνει αυτό, όταν κάποιος υποπτεύεται ότι κατηγορείται για κάτι, η δημιουργία του, το δικαίωμα θα πρέπει να δημιουργείται τη στιγμή που κάποιος είναι, γίνει ύποπτος για ένα δίκημα. Λοιπόν, τώρα έχει το λόγο ο κύριος Έντσιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία της και την εξαίρετη έκθεση που μας έχει υποβάλει. Να ευχαριστήσω όμως και την Επίτροπο Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ η οποία πρότεινε είναι την οδηγία. Η νέα ε, αυτή πρόταση οδηγίας ε, τελικά απαντά σε ένα πολύ σημαντικό ε, ερώτημα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε 27 χώρες μέλη. Ε, καταδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη μεγαλύτερης εναρμόνισης των νομικών και ποινικών συστημάτων. Το πρώτο βήμα στην διαδικασία αυτή είναι η κοινή και σωστή πληροφόρηση ε, του, του υπόπτου ή του κατηγορουμένου. Ε, σε μια γλώσσα που να κατανοεί και όχι απαραίτητα στη γλώσσα της χώρας στην οποία έχει συλληφθεί γιατί αυτό μπορεί να είναι κατάχρηση. Οι Ρωμά ας πούμε από τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία ε, διώχθησαν από την Γαλλία χωρίς να γνωρίζουν καν ε, το κατηγορητήριο γιατί δεν κατανοούσαν την γαλλική γλώσσα. Αυτή είναι παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελευταίος αγορητής είναι ο συνάδελφος κύριος Ζιόμπρο, ο οποίος θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το δικαίωμα της ενημέρωση στις ποινικέ διαδικασίες, ενημέρωση των υπόπτων για τις κατηγορίες που απαγγέλλονται εναντίον τους, πρέπει να είναι πρότυπο μια τυποποιημένη κατηγορία στα κράτη-μέλη. Ε, είναι λοιπόν πολύ σοβαρό που σε αυτό το σώμα μας απασχολεί το ζήτημα. Μας ακανοποιούν λοιπόν τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα συμπεριληφθούν στην οδηγία αυτή, αλλά δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να ξεχνάμε και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη, όπως το δικαίωμα των θυμάτων που πολύ συχνά βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και που δεν ενημερώνονται επειδή καθίστανται, ε, ε, παρότι είναι θύματα πολύ σκληρών και άγριων εγκλημάτων. Τέτοιου είδους εγκλήματα για τέτοια κλίματα κατηγορούνται σε χώρες τις οποίες είναι τουρίστες ή επισκέπτες και όπου δεν μπορούν να επισκεφθούν τον εαυτό τους για το λόγο γλωσσικών εμποδίων. Δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει δυσαναλογία μεταξύ θυμάτων και κατηγορουμένων. Μην ξεχνάμε ότι τα θύματα περνούν από μια δευτερογενή κατάσταση. Μιλάμε για δευτερογενή ε, δημιουργία θυμάτων. Δηλαδή ξαπεναπερνάνε τις δύσκολες καταστάσεις. Το κράτος πρέπει να τους φροντίζει. Πρέπει να τους ε, ε, παρασχεθεί φροντίδα. Ενώ οι εγκληματίες, οι οποίες πολύ συχνά συνεργάζονται σε ομάδες, χαίρουν μεγαλύτερης και καλύτερης υπεράσπισης από ό,τι τα θύματα. Θα πρέπει εδώ να υψώσουμε τη φωνή μας υπέρ αυτών των θυμάτων και θα ήθελα η Επίτροπος να δεσμευτεί, να εργαστεί για τα θύματα για αυτούς που έχουν δυστυχώς πέσει θύματα σε διάφορες, διαφορών καταστάσεων. Αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζιόμπρο. Τώρα τελειώσαμε το γύρο των αγορητών και θα περάσει στη διαδικασία catch ε, the eye. Καταρχήν έχει το λόγο για ένα λεπτό η κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ποινική νομοθεσία των κρατών μελών πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλα τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες της Ευρώπης. Η τροπολογία 4 αναφέρεται στο δικαίωμα για μετάφραση και διερμηνία. Αυτό είναι σε σαφής εφαρμογή της αρχής της πολυγλωσσίας που εμπεριέχεται στις ιδρυτικές συνθήκες και καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωμα για δωρεάν ε, δικηγόρο που η ίδια τροπολογία περιλαμβάνει αντικατοπτρίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο και την αρχή της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Τέλος, στο μέτρο, το μέτρο αυτό είναι σημαντικό για να γίνει σεβαστή μια βασική ελευθερία Είμαι υπέρ του γεγονότος ότι κάθε κρατούμενος ή ε, ε, συλλαμβανόμενος πρέπει να ε, λαμβάνει αυτό το έγγραφο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το ελάχιστο επίπεδο ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πασέσκου. Τώρα ο κύριος Πρέντερκαστ έχει το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Η δικαστική συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι όπως οι, κατηγορούμενοι ή οι εγκληματίες πρέπει να προσπαθούν να βρουν τρόπους για να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις ε, στα κράτη-μέλη, θα πρέπει και οι κατηγορούμενοι να μην ε, ε, υφίστανται συνέπειες διαφορών των δικαστικών συστημάτων. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα εξασφαλίσει ότι όταν κάποιος κρατείται ή συλλαμβάνεται στην στην Ευρώπη θα έχει την εγγύηση ενιαίας ε, διαδικασία. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι αυτοί που κρατούνται στις επικράτειές τους θα ενημερώνονται παρκώς για τα δικαιώματά τους. Παρότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν προσυπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξακολουθούν να παραβιάζονται τα ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη που έχουν τα δικαστικά συστήματα μεταξύ τους και αυτό μπορεί να ισχύσει όταν όλα τα, όσα ισχύουν στην Ευρώπη είναι παντού τα ίδια. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Εάν ένας πολίτης διαφορετικής ε, χώρας βρεθεί σε μια ε, δυσχερή κατάσταση σε μια άλλη χώρα όπου δηλαδή βρίσκεται υποπτωσή κατηγορούμενος τότε αυτός φαίνεται ότι βρίσκεται σε απελπισμένη κατάσταση γιατί πραγματικά τις περισσότερες φορές δεν ξέρει τι τον περιμένει, τι πρέπει να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η νέα οδηγία είναι πολλά υποσχόμενο και θετικό σημάδι ε, ότι υπάρχει μια αρχή κοινών ε, ε, προτύπων ε, που θα ισχύσουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές να μην υποπέπτουν, υποπίπτουν διαρκώς σε λάθη και από την άλλη πλευρά να μπορούν να ασκήσουν καλά την δράση τους, σωστά τη δράση τους. Θα βελτιωθεί με τον τρόπο αυτό η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπάλτσερ. Ναι, κατ' ουσία θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και σε υπεράσπιση θα πρέπει να εδραιώνεται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η ενημέρωση των κρατουμένων δεν παρουσιάζει προβλήματα. Ωστόσο, ε, υπάρχουν ετησίω 8 εκατομμύρια υποθέσεις όπου δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση των κρατουμένων και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε μια άλλη χώρα δεν μπορούν να ενημερωθούν σε μια γλώσσα που κατανοούν για τα δικαιώματά τους. Σε ορισμένες χώρες η ενημέρωση γίνεται προφορικά, σε άλλες γίνεται γραπτά, αλλά σε μια τόσο πολύπλοκη γραφειοκρατική ξύλινη γλώσσα που ακόμα και στη μητρική γλώσσα χωρίς να έχει κανείς νομικές γνώσεις δεν μπορεί να την καταλάβει. Θα πρέπει λοιπόν να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι τώρα θα γίνεται γραπτά η ενημέρωση των ε, κατηγορουμένων με έναν εύληπτο τρόπο ε, ούτως ώστε να μπορεί το απλό αυτό μέτρο να είναι χρήσιμο για την αποφυγή των δικαστικών πλανών. Η τελευταία παρέμβαση είναι η παρέμβαση της κυρίας Σίγκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα εκπλαγούν πολύ από την εκλογική μου περιφέρεια όταν ακούσουν αυτά τα δικαιώματα που θα έχουν τώρα. Ενδεχομένως βέβαια θα, αναγνωριστούν, θα αναλογιστούν ε, σε ποια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος ε, η χώρα τους. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει το ευρωπαϊκό ε, ε, έντυπο έκδοσης το οποίο μπορεί να επιτρέψει σε άλλες χώρες να συλλάβουν ή να, εκδώσουν έναν Βρετανό υπήκο. Θα πρέπει να διαλέξουμε τι είδους Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε. Ολοκληρώσαμε το κύριο Catch και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην ε, Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, η οποία θα απαντήσει σε όλες τις παρεμβάσεις. Έχετε το λόγο κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σπάνια περίπτωση στο θεσμικό αυτό όργανο όλες οι πολιτικές ομάδες από, την τη δεξιά προς την αριστερά και του κέντρου συμπεριλαμβανομένου να συμφωνούν ε, σε ένα μέτρο. Και μοιάζει ότι εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που αύριο... Αυτό το οποίο συνέβη στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα επαναληφθεί. Μια συντριπτική πλειοψηφία θα υποστηρίξει την απόφαση αυτή. Και όσο ταχύτερα εφαρμοστεί και τεθεί η ισχύ αυτή η οδηγία, τόσο το καλύτερο. Φυσικά, μιλάμε για την πλήρη ε, μεταφορά της στο δίκαιο των κρατών μελών, που και αυτή πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Αυτό θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη σοβαρολογεί όταν μιλά για προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ότι περισσότεροι από εσά που πήρατε σήμερα το λόγο ήδη εργάζεστε για το τρίτο μέτρο του οδικού χάρτη ε, των ε, δικονομικών δικαιωμάτων της πρόσβασης σε δικηγόρο. σε δικηγόρο. Είμαι πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει την Επιτροπή στο θέμα αυτό, διότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία πραγματικά αντιδρούν στην παρουσία δικηγόρου και υπολογίζω στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να επέλθει μια σωστή ισορροπία στην πρόταση αυτή ανάμεσα στο δικαίωμα της υπεράσπισης και στο, στην ανάγκη να γίνουν αποτελεσματικά οι ποινικέ ε, έρευνες. Ε, αισθάνομαι πολύ καλύτερα που βρίσκομαι στα χέρια του Κοινοβουλίου για τη βελτίωση ενός ε, κειμένου το οποίο πρέπει να υπάρξει. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε αυτό, ευχαριστώ που θα το υπερψηφίσετε αύριο και σας ευχαριστώ που θα μας βοηθήσετε στα επόμενα μας βήματα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Η ομοφωνία στην οποία αναφερθήκατε είναι ο καλύτερος τρόπος για να συγχαρούμε την Επιτροπή για το έργο της. Τώρα θα κλείσουμε τη συζήτηση δίνοντα το λόγο στην συγκίτρια την κυρία Ζίπελ, η οποία έχει δύο λεπτά για την τελική της παρέμβαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ε, στην αρχή μίλησα υπερβολικά αργά και γι' αυτό ξεπέρασα το χρόνο μου. Γι' αυτό θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Η κυρία Ρέντινγκ είπε ότι η συζήτηση σήμερα τόνισε αυτό που έδειξε η ομόφωνη απόφαση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Δηλαδή ότι η ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων είναι ένα κοινό ενδιαφέρον όλων των πολιτικών ομάδων. Γι' αυτό έχω την πεποίθηση ότι και το επόμενο μέτρο, το δικαίωμα της ε, προσφυγής σε δικηγόρο θα, δημιουργήσουμε, θα έχουμε μια καλή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία θα μπορέσουμε εμείς να τη βελτιώσουμε περαιτέρω και στη συζήτηση με το Συμβούλιο θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή οδηγία. Θα ήθελα να ευχηθώ εδώ στην εισηγήτρια κυρία Αντανέσκου καλή επιτυχία και να της πω ότι μπορεί πραγματικά να υπολογίζει στη σύρρηξη του σώματος. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ζήπελ. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που εξοικονομήσετε χρόνο. Ε, κλείνει λοιπόν εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Τώρα θα περάσουμε στα επόμενα